Καλημέρα. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν συμφωνούμε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ωραία. Και προχωρούμε στο δεύτερο σημείο Στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης θα παρουσιάσουμε την ε, ενδιάμεση έκθεση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, Εκρίζωσης ε, της Εμπορίας Ανθρώπων. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελευθεριών. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, τον κύριο Μωράες, Πιστεύουμε ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η κοινή συνάντηση. Έχουμε μαζί μας ε, την κυρία Βασιλάδου, Βασιλιάδου, συγγνώμη, ε, που είναι η Ευρωπαία Συντονίστρια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ε, είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ ε, των κρατικών πολιτικών, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δράσεων των διαφορών υπηρεσιών και οργανισμών. 18 Οκτωβρίου ήταν η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων και η Κομισιόν με αυτή την ευκαιρία υπέβαλε αυτή την ενδιάμεση έκθεση την οποία θα σχολιάσουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Βασιλιάδου για την παρουσία της σήμερα και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελευθεριών, τον κύριο Μωρές. Thank you very much, um, Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ε, οργάνωση αυτής της ανταλλαγής απόψεων, αυτής της συζήτησης σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Δεν είναι καινούριο θέμα, ξέρουμε τη σημασία του. Αρχίσαμε τη συζήτηση στην τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου με την υιοθέτηση της οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων που είναι η πρώτη οδηγία ε, ε, νομικής φύσεως και ε, ποινικού δικαίου που υιοθετήθηκε από αυτήν την Επιτροπή ένα από τα στοιχεία ήταν ορισμός ε, ενός ε, συντονιστή μια συντονίστρια ε, για την διαμόρφωση της πολιτικής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Είναι συντονίστρια λοιπόν δράσης. Είναι μια, ένα γεγονός το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα διότι άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάζει τα σεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και έχει πάρα πολλές περίπλοκες, περιπλοκές και παράπλευρες επιπτώσεις. Περιμένουμε λοιπόν ε, με μεγάλη χαρά την παρουσίαση της εκθέσεως της συντονίστριας σήμερα. Μάλιστα είχαμε μία πρόσφατη έκθεση η οποία έδειξε πως έχει ανέβει το ποσοστό της, ε, ε, των σκλαβωμένων ανθρώπων σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να δώσω απευθείας το λόγο στην κυρία Βασιλιάδου Είναι, Είμαι, πάρα πολύ τυπικό σήμερα και εξαιρετικά ευγενής, αλλά καλό είναι να προχωρήσουμε κατευθείαν με την συντονίστρια, την κυρία Βασιλιάδου. 20 λεπτά. Στην Επιτροπή ε, Λίμπε δίνουμε χρόνο, 20 λεπτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω την ε, πολιτική ε, της καταπολέμησης της εξάλληψης εμπορίας ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έχετε υποστηρίξει σημαντικότητα στο δύσκολο έργο μου και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έχουμε ένα περίπλοκο πολιτικό και νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλο το δίκτυο της ε, συν, ε, Ο Επίτροπος κ. Αβρομόπουλος, εξέφρασε τη δέσμευσή του έναντι αυτού του θέματος και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει ε, να προβάλλει το θέμα αυτό της καταπολέμησης της εμπορίας των ανθρώπων ως μια προτεραιότητα του ντοσχέτου. Η εμπορία ανθρώπων ε, αντιπροσωπεύει μία τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι μία ε, μεγάλη σημαντική πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι μία μορφή του οργανωμένου εγκλήματος που απαγορεύεται συγκεκριμένα, αναφέρεται δηλαδή στον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Όταν λοιπόν καταπολεμούμε εμπορία ανθρώπων, ε, εφαρμόζουμε τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα όμως, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που μεμονωμένα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνα τους και γι' αυτό πρέπει να συντονίσουμε και να οργανώσουμε την, τον αγώνα μας, τις δράσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως ήδη συζητήθηκε, ε, έχει, έχω ήδη πει δηλαδή, θα σας ε, αναφέρω τι συζητήθηκε το 14 Οκτωβρίου, η οποία ήταν η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά της ανθρώπινης εμπορίας, εμπορίας ανθρώπων. Είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τηρούνται, είναι δέσμοι και δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν ουσιαστικά σκλαβωμένοι και υποχρεώνονται με το ζόρι να εργαστούν. Ε, είναι, έχουμε εντοπίσει διάφορα τέτοια κυκλώματα και ακούμε φρικιαστικές ιστορίες ε, ανθρώπων που ε, είναι εγκλωβισμένοι δίπλα μας και δεν είχαμε πάρει είδηση. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μακριά και απομονωμένα, αλλά για να σας δώσω μια ιδέα, μεταξύ του 2010 και 2012, 30, 146, 30.146 άνθρωποι, γυναίκες, άνδρες, παιδιά, είχαν καταχωρηθεί ως εγκλωβισμένοι σε, ουσιαστικά σε σκλάβοι δηλαδή, ως εργαζόμενοι με τη βία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η, η, επίσημη κατα, ε, καταχωρημένη ως ε, ως εγκλωβισμένοι ε, σε, εργασία διά της βίας. Πολλές φορές είναι γυναίκες οι οποίοι διακινούνται από σωματέμπορους και αναγκάζονται να εκδοθούν. Άλλες φορές είναι οικιακές ε, ε, βοηθοί, δηλαδή γυναίκες οι οποίες με το ζόρι υπηρετούν σε σπίτια χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα και άλλες φορές είναι και άντρες σε οικοδομές ή σε άλλα επαγγέλματα. 80%, 80 των σημάτων είναι γυναίκες, 70% των, ε, των, διακινητών είναι άντρες και 16% των σημάτων είναι παιδιά. Ε, το 69%, ε, το 69% συντριπτικό ποσό είναι γυναίκες οι οποίες εργάζονται ως ιερόδουλες, γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Χίλια παιδιά ε, ανακαλύφθηκαν ότι διακινούνταν από διακινητές για σεξουαλικούς λόγους. Σεξουαλική εκμετάλλευση. Αλλά δεν είναι μόνο αποκλειστικά γυναίκες και κορίτσια. Είναι και άντρες και αγόρια. 67% των θυμάτων προέρχονται από χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Ουγγαρία και Πολωνία. 67% και τα υπόλοιπο ποσοστό των θυμάτων είναι από την Ιγυρία, Βραζιλία, Κίνα, Βιετνάμ και Ρωσία. Οπότε οι περισσότεροι εγκληματίες ε, διακινητές και τα περισσότερα σήματα είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Και γιατί το τονίζω αυτό. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε την ε, εμπορία ανθρώπων και την ε, παράνομη διακίνηση ως ταυτόσιμες έννοιες. Υπάρχουν όμως υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία ξεχωρίζει σαφέστατα τους λάθρομετανάστες, αυτούς που εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο νομικό πλαίσιο που καλύπτει την εμπορία ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι εισέρχονται λαθρέ εν συνεχεία ε, εγκλωβίζονται και διακινούνται για σεξουαλικούς λόγους ή ε, ε, σκλαβωμένη εργασία. Είναι λοιπόν ε, παρήγορο από τη μία πλευρά ότι έχουμε μία σωστή νομική βάση που μας διευκολύνει να αναλύουμε σωστά τα δεδομένα που έρχονται στα χέρια μας. Τώρα δεν είναι μόνο τα, τα ορισμός ε, που, που των ανθρώπων αυτών που είναι μεγάλος, 10, 20, 30 χιλιάδες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι και η πραγματικότητα της ζωής που ζούνε. Πρέπει να επικεντρωθούμε και στο ποινικό δίκαιο, στις ε, προσφυγές τους και στα δικαιώματά τους ως άνθρωποι. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να είμαι σαφέστατη. Είναι πάρα πολύ ωραία το ρόλος μου ως συντονίστριας να συμβουλεύω και να διαβουλεύουμε με τα, τους ενδιαφερόμενους ε, φορείς. Αλλά δεν είναι αυτό το έργο μου, το εγώ ε, επιτελώ μια, ε, μια εργασία που έχει νομική υποχρέωση. ο νόμος με υποχρεώνει, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με υποχρεώνει να κάνω τη δουλειά μου αυτή η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 23 της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ε, όσον αφορά λοιπόν την νομοθεσία, το νομοθετικό μας πλαίσιο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο που υποτίθεται θα, θα μεταφέρεται στις 6 Απριλίου του 2013 σε όλα ε, τα δίκαια, την νομοθεσία των κρατών μελών. 25 ε, κράτη-μέλη πλην της Γερμανίας και του Βελγίου, 25 λοιπόν έχουν μεταφέρει τη διατάξη οδηγίας στην εθνική του νομοθεσία, εκκρεμεί ακόμα στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Δεν θα, θα, επιβάλλουμε την αναγκαία πίεση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς και σε αυτές τις δύο χώρες. Έχουμε λοιπόν μία σαφή υποχρέωση να υποστηρίζουμε ε, τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή αυτής της ε, νομοθεσίας, της οδηγίας και η στρατηγική μας ήταν εξαιρετικά συνεπής, ολοκληρωμένη ε, και το ήταν το αποτέλεσμα πάρα πολλών ε, ενδιαφερομένων και θυγόμενων πλευρών. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που ε, ενδιαφέρονται και θέλουν να εφαρμόσουν ε, τα συμπεράσματα του, Συμβουλίου και η στρατηγική αυτή έχει επιπτώσει σε ολόκληρη την Ένωση. Η ενδιάμεση λοιπόν έκθεση παρουσιάζει τα επιτεύγματά μας μέχρι σήμερα με τη συνεργασία της, των κρατών μελών, των ε, αρμοδίων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών και της διευθύνσης της Κομισιόν, αλλά και με χώρες που εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν καταγράψει τα πεπραγμένα, είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για την εργασία μας, διότι εγκαίρως παρουσιάσαμε την έκθεσή μας και πιστεύω ότι τηρήσαμε όλες μας τις υποχρεώσεις και υποσχέσεις τονίζω ορισμένες πτυχές της εργασίας μας η συνέχιση της των αναφορών που λαμβάνουμε μέσω των διαφόρων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δηλαδή τώρα τα κράτη-μέλη συνεργάζονται πολύ στενά με την Κομισιόν. Έχουμε δημιουργήσει μία πλατφόρμα ε, με πάνω από 100 μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ναι, οι οποίες συνεργάζονται ε, για να παρακολουθούν και να ανταλλάσσουν απόψεις για την κατάσταση της εμπορίας και μπορούμε εμείς τώρα να είμαστε σε επαφή και να ενημερωνόμαστε αλλά και να ενημερώνουμε το τι συμβαίνει σε αυτό τον τομέα. Μαθαίνουμε από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μαθαίνουμε τι εργασία επιτελούν και τι εμπειρίες έχουν. Και αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ε, επίτευγμα. Έχουμε επίσης ξεκινήσει μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα ε, με την οποία θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, εμπειρίες και όλα αυτά τα στοιχεία ιδραίων στην έκθεσή μας. Έχουμε δημοσιεύσει εγχειρίδια, ενημερωτικά φυλάδια για το πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τα σήματα, να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά τους, να προφυλάξουμε παιδιά και σε άλλα πολλά θέματα. Έχουμε επίσης ε, ξεκινήσει μελέτες για ε, ευάλωτες ομάδες, νομολογία ε, και άλλα θέματα. Κατά την ημερίδα λοιπόν της ε, Ευρώπης για κατά της εμπορίας έχουμε, παρουσιάσαμε την ενδιάμεση έκθεση, την έκθεση της Eurostat και το τρίτο στοιχείο του πακέτου ήταν η δεύτερη έκθεση υλοποίησης για τις προσωρινές άδειες παραμονής ε, ε, ε, ατόμων που έχουν εισαγένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσετε τα συμπεράσματα της έκθεσης, διότι δυστυχώς αυτό που είδαμε, ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται στο 100% του δυναμικού της από όλα τα κράτη-μέλη. τώρα, σε τι ε, σημεία εστιάζουμε. Καταρχάς τα παιδιά. Έχουμε ταυτοποιήσει ποια παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα για εμπορία ανθρώπων είναι ένας ε, φαύλος κύκλος της εμπορίας παιδιών και ένας από τους, ε, από τους στόχους μας ε, το, του 2014 ήταν να δημοσιεύσουμε μαζί με τον υπηρεσία του ΟΗΕ ένα χειρίδιο που να αναφέρει όλες αυτές τις πτυχές της εμπορίας παιδιών. Έχουμε ξεκινήσει και διάφορες δράσεις θα μου πείτε τώρα ότι 16, μόνο 16% των ταυτοποιημένων σημάτων είναι παιδιά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία το ποσοστό. Πρέπει να κάνουμε το έργο μας σωστά και να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τα δίκτυα προστασίας των παιδιών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, διευρύνουμε την ενομέρωση, προσφέρουμε συμβουλές ε, και ολοκληρώνουμε όλο αυτό το δίκτυο προστασίας το 2015. Όσον αφορά τώρα τη διάσταση των φύλων, ε, όχι, θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό, όχι μόνο επειδή είμαι ενώπιον της Επιτροπής για τη Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, αλλά επειδή και αυτό αποτελεί μια πτυχή του έργου μας και το, ε, τονίζει, το τονίζουμε. Επανέρχομαι λοιπόν στο συνέδριο του ΟΗΕ πριν από δύο χρόνια για τις γυναίκες και το οποίο αναγνώρισε στα συμπεράσματα ότι η διακίνηση γυναικών είναι ακριβώς ε, ε, ε, μια πτυχή της εμπορίας ατόμων. Βασικά η εκμετάλλευση των γενικών οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα, σεξουαλική διακίνηση, σεξουαλική εκμετάλλευση και πολλά άλλα φρικιαστικά. Ε, είναι Λοιπόν και αυτό ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα διότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αυτά που διακινούνται και είναι σήματα γίνονται εξαιρετικά ευάλωτα και πρέπει να προσφέρουμε ένα δίκτυο στήριξης και προστασίας. Το βασικό, βασικά είναι σήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης όπως έδειξε και η έκθεση του Eurostat. Πορνεία, ε, σε ιδιωτικό χώρο, έξεση σε δημόσιους χώρους όπως γίνεται σε διάφορες περιοχές, ε, ιερόδουλες, ε, όλες τις, όλο των ειδών της σεξουαλικής, εμπορίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά εμπορίας γυναικών η οποία έχει άμεση σχέση με την πορνεία και την παροχή των γυναικών αυτών σε, για πορνεία και εκμετάλλευση. Είναι ένας τομέας αυτός ο οποίος πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και διονγκώνεται διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ε, προτάσεις ε, του Κοινοβουλίου για την προστασία γυναικών από σεξουαλική εκμετάλλευση. Έχουμε, ε, διαβα... έχουμε, ακολουθούμε τις συστάσεις της έκθεσης και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, την εφαρμόσουμε. Η έκθεση αυτή περιλάμβανε και την ε, προοπτική, της, την πτυχή της πορνείας. Η σεξουαλική ε, εκμετάλλευση είναι ε, ε, έγκλημα ευρωπαϊκού επίπεδου. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει συγκεκριμένα την σεξουαλική εκμετάλλευση και βάσει της οδηγίας 2011 ε, δεν περιλαμβάνει την σεξουαλική εκμετάλλευση. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν μιλάω λοιπόν για εμπορία ατόμων για σεξουαλική ε, εκμετάλλευση, μιλώ συγκεκριμένα για την εμπορία και τη διακίνηση των γυναικών και κοριτσιών αυτών. Θέλω και συνέχεια τονίζω αυτό το πρόβλημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όχι όμως μόνο από τη γυναική πλευρά, αλλά και από την πλευρά των ανδρών και αγοριών. Τα παράλληλα με την εκμετάλλευση για εργασία, δια της βίας. Αυτά τα άτομα ε, πρέπει να προστατευθούν, πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αρχές να μπορούν να καταγγείλουν Γι' αυτό ε, επειδή λοιπόν είναι δυσανάλογο το ποσοστό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης εστιάζουμε πάρα πολύ στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Πρώτο λοιπόν θέμα εστίασης ήταν αυτό. Δεύτερο νομολογία. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε το νομικό υπόβαθρο, θέλουμε να ε, προστατεύσουμε όλα τα θύματα. Το ότι δεν καταγράφονται τα θύματα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι είναι σκλαβωμένοι σε, στα σπίτια και προσφέρουν οικιακές υπηρεσίες με διαβίας. Υπάρχουν άνθρωποι των, των οποίων ε, είναι σήματα διακίνησης οργάνων για μεταμοσχεύσεις και άλλες πολλές μορφές. Είναι δηλαδή η αγοραπολισία ανθρώπων και ε, των υπηρεσιών που προσφέρουν οι άνθρωποι αγοραπολισία ανθρώπων, οργάνων ανθρώπων. Λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ευάλωτοι διότι στις πατρίδες τους ε, υπάρχουν, γίνονται σειράξεις, πόλεμοι, υπάρχει ανισότητα. Εγώ διαφωνώ, δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος. Υπάρχει τρομερή, τρομακτική φτώχεια στον κόσμο και αυτή η εμπορία υπάρχει, γίνεται, πρώτον επειδή είναι πολύ προσοδοφόρα και δεύτερον επειδή υπάρχουν τα, υπάρχουν τα, οι ευάλωτες αυτές ομάδες του πληθυσμού, τα θύματα. Αυτό το αναγνωρίζει και η Europol στην έκθεσή της του 2013 που λέει ότι αυξάνεται η ζήτηση για διακίνηση πίσω από κάποιο θύμα υπάρχει ένας εγκληματίας, ένας διακινητής και υπάρχει και κάποιος που θέλει τις υπηρεσίε του θύματος. Μιλάμε για 200 δισεκατομμύρια κέρδος ευρώ ε, παγκοσμίω. Ένα τεράστιο τέτοιο ποσό που αντιπροσωπεύει το κέρ, τα κέρδη. Αυτά, ε, αυτά τα δισεκατομμύρια τα αποφελούνται οι διακινητές. Ε, αλλά ε, τα εποφελούνται και διάφοροι νομικοί, τα διάφορα δίκτυα δικηγόρων, νομικών, οι οποίοι προσπαθούν πολλές φορές να μας, ε, κλείσουν, να μας κουκουλώνουν τα εγκλήματα, προσπαθούν να μας κλείσουν τα μάτια κλπ. Αλλά ε, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Όλοι αυτοί και οι διακινητές και οι δικηγόροι τους και οι... αυτοί που θέλουν τις υπηρεσίες ε, των θυμάτων είναι Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι πολίτες. Τονίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά και με αυτούς που προσπαθούν να διασφαλίσουν την ε, ασφάλεια του κυβερνοχώρου, διότι υπάρχουν και πολλά υπόγεια ρεύματα στον κυβερνοχώρο, τα οποία διευκολύνουν αυτές τις δραστηριότητες. Όσον αφορά τώρα τη ζήτηση ε, για τις υπηρεσίες μας, εγώ δεν συμβουλεύω τους ανθρώπους απλώς λέγοντας ή τους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να μειώσουμε την ζήτηση για, την, ε, ε, για τις εγκληματικές αυτές ε, πράξεις. Όχι, το λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει μαζί με την καταπολέμηση του φαινομένου πρέπει να καταπολεμηθεί και η ζήτηση. Δηλαδή να καταπολεμήσουμε αυτούς τους οποίοι, οι οποίοι επιζητούν τις υπηρεσίες των διακινουμένων και να τιμωρηθούν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταστήσουμε σαφές ότι ένα έγκλημα είναι ποινικό. Πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτό αυτό και σας ρωτώ, ξέρουμε άλλες εγκληματικές ενέργειες που δεν υπάρχουν ποινικέ επιπτώσεις, δεν θεωρείται δηλαδή εγκληματίας αυτός ο οποίος διαπράττει το έγκλημα, την αδικοπραξία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου και την ε, οδηγία για, την, για κυρώσεις κατά των εργοδοτών του 2009 ε, η οποία ε, λέει ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν όσοι απασχολούν θύματα εμπορίας ε, ανθρώπων. Δηλαδή ένας εργοδότης ο οποίος ξέρει ότι εσύ έχεις υπάρξει θύμα και σε προσλαμβάνει πρέπει να τιμωρηθεί βάσει των διατάξεων που έχουν ψηφιστεί. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να συνεργαστούμε με το δημόσιο ιδιωτικό τομέα, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πρέπει να συνεργαστούμε με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε και μία έκθεση για τις δράσεις τις οποίες ε, κάνουμε. Έχουμε ορισμένες χώρες προτεραιότητος για συνεργασία. Ουκρανία, Βραζιλία, οι χώρες του, της ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης και αυτές είναι εξωτερικές μας ε, δράσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι αντιπροσωπείες μας. Λοιπόν, δουλεύουμε για την προστασία των θυμάτων, για τον εντοπισμό των θυμάτων, ε, συνεργαζόμαστε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζουμε τις διατάξεις της οδηγίας, ε, σύμφωνα με το άρθρο 20 πάλι που διαγράφει το, το, το, περιεχόμενο της εργασίας μας θα συντάξουμε μία έκθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και το την έκθεση αυτή την θα την υποβάλλω στην Κομισιόν και η τελευταία έκθεση είναι βασισμένη στο άρθρο 23 ε, για την ποινικοποίηση του αδικήματος. Ε, όλες αυτές τις εκθέσεις λοιπόν τις υποβάλλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπερασματικά πρέπει να ε, πω ότι έχουμε την ομοθεσία, έχουμε την νομική βάση, έχουμε την πολιτική την οποία εφαρμόζουμε, έχουμε και πιστώσεις, έχουμε τα κονδύλια και τα κονδύλια αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Αυτά όλα τα έχουμε, αλλά αυτό που δεν έχουμε είναι πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και πλήρη εφαρμογή του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου. Ε, ότου λοιπόν ε, ε, εφαρμόσουμε 100% όλο το νομικό δίκτυο που υπάρχει στη διάθεσή μας και όλες τις ε, διατάξεις θα έχουμε αποτύχει έναντι των πολιτών και των κοινωνιών μας. Διότι ε, στο κάτω-κάτω της γραφής ε, πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και να μην τους προσβάλλουμε, να μην δεχόμαστε ότι ξαφανίζονται, δολοφονούνται, σκοτώνονται, βιάζονται ε, και κάθε λεπτό που περνάει είναι πολύτιμο για τη ζωή τους. Ευχαριστώ. Eh, eh, Ευχαριστώ κυρία Βασιλιάδου. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας στην Επιτροπή. Είπατε πολλά σημαντικά. Που είναι και πολύ χρήσιμα για τις Επιτροπές μας. Αρχίζει η συζήτηση. Έχουν δηλώσει πολλοί ότι θέλουν να λάβουν το λόγο. Δεν μπορώ να δώσω στον καθένα πάνω από δύο λεπτά μέγιστο χρόνο. Η κυρία Χέρτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε και πάλι. Ελπίζω ότι θα σας συναντούμε συχνότερα στο μέλλον, γιατί το θέμα της εμπορίας ανθρώπων είναι πολύ μεγάλο. Δύο ερωτήσεις. Ε, η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση για την εμπορία ανθρώπων και λέει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες πλήττονται με διαφορετικό τρόπο. Οι δε στατιστικές δείχνουν ότι κυρίως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών αυξάνεται, όπως είπατε κι εσείς. Η φετινή χρονιά από τη Europol και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε αναφορά μεταξύ υποχρεωτικής ε, πορνείας και εμπορίας ανθρώπων. Τι συμπεράσματα ε, μπορούμε να εξαγάγουμε από εδώ. Επίσης είπατε ότι τώρα τρέχει μια μελέτη που θέλει να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και θα δημοσιευτεί αρκετά σύντομα, δηλαδή το πρώτο εξάμεινο του 2015. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, έχει το Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω ότι υποστηρίζω απόλυτα αυτά που μας είπατε για τις διαφορές που υπάρχουν πολλές φορές μεταξύ των λαθρεμπόρων και της εμπορίας, η διακίνησης. Αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική και εδώ και αλλού όταν χρησιμοποιούμε ως συνώνυμα τις δύο λέξεις. Προκειμένου περί των διαφορετικών μορφών εμπορίας διακίνησης και των διαφορετικών ε, ε, τομέων, είτε είναι πορνεία ή ένα σωρό ε, τομείς που κι εσείς αναφέρατε. Αναρωτιέμαι τι κάνουν στην πραγματικότητα τα κράτη-μέλη μας και αν όντως έχουν εμπλακεί ενεργά για να καταπολεμήσουν κάποιες μορφές εμπορίας. Διότι πάντα υπάρχουν ε, άνθρωποι που γνωρίζουν, υπάρχουν ειδικοί, μπορεί κάποιος, μπορεί, ε, κάποιος που εργάζεται σε ένα αρτοπείο να μην δίνει στόχος ε, ε όμως ο εκδιοκτήτης γνωρίζει γιατί ε, αν τον πληρώνει, τον πληρώνει λίγο, δεν πληρώνει ε, ασφαλιστικές φορές κλπ. Οπότε βγάζουν κέρδος και έχουμε την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη δεν καταπολεμούν ενεργά τέτοιου είδους μορφές εκμετάλλευσης και επίσης στον τομέα της πορνείας. Τι πιστεύετε, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αποτελεσματικές μορφές καταπολέμησης αυτών των ε, μορφών εκμετάλλευσης και υπάρχουν διαφορές αντιμετώπισης ε, μεταξύ κρατών μελών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θέλω να κάνω μια-δυο ερωτήσεις. Πρώτον, θέλω να ξέρω ποιο ποσοστό αυτών των πολλών νέων ανθρώπων, ε, αγοριών και κοριτσιών, απάγονται και σε ποιο βαθμό υπάρχει ε, η θελημένη εμπορία, όχι ότι οι ίδιοι θέλουν να γίνουν αντικείμενα εμπορίας, αλλά μπορεί να τους έδωσαν οι γονείς ή οι συγγενείς. Καμιά φορά ένας λόγος αποχωρισμού των αγαπημένων προσώπων θα έλεγα, ε, ποιος, λόγος είναι αυτός. πολλέ πολλές φορές υπάρχει κάποιος λόγος. Γιατί τους πουλούν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. κυρία Ιμπέρ. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για την έκθεση. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, αν μια χώρα δεν θέλει να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, όπως τη Σουηδία, τη δική μου τη χώρα, αν δεν αφήνει τους συνοριοφύλακες να κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων. Σε ποιο βαθμό αυτό αυξάνει την εμπορία ανθρώπων. Δεύτερον, είπατε ότι αυξάνεται η επαιτία και ο αριθμός των επαιτών στους δρόμους της Ευρώπης. Και αυτό είναι μορφή εμπορίας, είπατε. Πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Μπορεί ε, ε, ε, γιατί στη Σουηδία επισήμως ε, αρνούνται την ύπαρξη επετών. Αυτή η επίσημη πολιτική μπορεί ίσως να επιδεινώσει το πρόβλημα της επαιτίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόζεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Βασιλιάδου, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πολύ αναλυτική και στατιστική καταμέτρηση των συμπτωμάτων της εμπορίας, δηλαδή ανθρώπων και οργάνων, όπως εξειδικεύσατε, ειδικά αναφερόμενοι στην κατηγορία των ανήλικων παιδιών. Εδώ α, ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση. Σωστά είπατε ότι είναι πολλοί εκείνοι που εμπλέκονται σε αξιόπινες πράξεις σχετικά με την εμπορία ανθρώπων. Υπάρχει προσφορά, υπάρχει και ζήτηση. Αλλά πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν ότι Παραδείγματο χάρη, ένα γιατρό που παίρνει μια εντολή να προβεί σε ένα χειρουργείο και να αφαιρέσει όργανα από ένα παιδί, προκειμένου αυτά τα όργανα να χρησιμοποιηθούν για εμπορική εκμετάλλευση. Είναι και αυτό απειλείται με κάθυρξη. Δηλαδή διαπράττει μια αξιόπινη πράξη, διότι προηγουμένω πρέπει να ελέγξει γιατί αυτό το παιδί, παραδείγματο χάρη, βρίσκεται στο χειρουργικό κρεβάτι και του αφαιρείται ένα νεφρό. Μιλάω για μια συνήθεια εμπορία οργάνων, που είναι η κατηγορία των νεφρών. Έχω ασχοληθεί και προσωπικά επαγγελματικά στην πατρίδα μου με μια τέτοια υπόθεση. Ε, σε κάθε περίπτωση σωστά επισημάνατε ότι ενδεχομένως από κράτος μέλος σε κράτος μέλος να διαφέρει η εφαρμογή της νομοθεσίας και ενδεχομένως και στην κατηγορία της πρόληψης να μην υπάρχει σωστή ενημέρωση, καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τη διάσταση, με πόσες περιπτώσεις περιλαμβάνονται στην κατηγορία εμπορία ανθρώπων και ποια είναι η ποινική πρόβληψη και ποινική μεταχείριση των δραστών που εμπλέκονται γιατί μιλάμε για διασυνοριακό έγκλημα, για εγκληματικές οργανώσεις που πλέον καλύπτουν όλο τον πλανήτη, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει και διασυνοριακή συνεργασία για όποια κατεύθυνση θετική, τουλάχιστον στις επιτροπές τις δικές μας και τη ΦΑΜ και τη ΛΥΜΠΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το αντικείμενο είναι, έχει προτεραιότητα και σε συνεργασία μαζί σας πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της πενταετίας μπορούμε να συμβάλλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μας ε, θυμήσατε δραματικά φαινόμενα που δείχνουν ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν απαραίτητος με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και θρησκευτικέ, ε, με την κοινωνία των πολιτών, να συνεργαστούν με εκείνους που καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με τα δεινά των ανθρώπων. Αυτό ε, αφορά ανθρώπους, μην το ξεχνάμε. στις πόλεις μας, ε, στους δρόμους μας, στις γειτονιές μας. Θα πρέπει να αναλυθεί η δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας και των δεινών των ανθρώπων. Είναι μια σύγχρονη δουλεία όλα αυτά. Δουλεμπόριο. Που παραβιάζει κατάφορα την νομοθεσία μας και πρέπει να τιμωρείται. Είπατε ότι 16% είναι παιδιά από τα θύματα των, ε, της εμπορίας ανθρώπων και σε ένα πρόσφατο σεμινάριο στα πλαίσια του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων αναφέρθηκε ότι αυτά τα παιδιά πολλούνται ε, και τιμώνται 40.000 ευρώ. Αυτό είναι κάτι που έχει τις πλέον διαφορετικές ρίζες και αίτια. Ε, πρέπει να δούμε και τη στάση την καταναλωτική τάση που σημειώνεται σήμερα, ε, εμπορία οργάνων κλπ. Επίσης ε, υπάρχει πορνογραφία, υπάρχει, υπάρχουν νέες ανάγκες γυναικών να γίνουν μητέρες με διάφορους τρόπους εμείς έχουμε και ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου που υπησέρχεται σε πολλά από αυτά τα θέματα και που συνάδουν με αυτά που μας είπατε κι εσείς. Και σας ευχαριστώ που μας τα είπατε όλα αυτά. Τέλος, να προσθέσω άλλη μια φορά ότι θα εξακολουθήσουμε να στηρίζομαι τις κατατόπους οργανώσεις που ε, εργάζονται σε αυτό το τομέα. Ε, Κλείνω τον κατάλογο των παρεμβάσεων. Απομένουν οκτώ άτομα ε, και πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο θέμα της Μέσιας διάταξης. Ο λόγος στην κυρία Σπινέλη. Όχι, όχι, ευχαριστώ κυρία Βασιλιάδου για την πολύ καλή παρουσίαση θα ήθελα να εκφράσω μια μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τη μη εφαρμογή των αντίστοιχων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια χώρα που την ξέρω καλά, την Ιταλία. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μελέτη του Ινστιτούτου Νομικών Μελετών σχετικά με τις διαφορετικές μορφές καταστρατήγησης των ευρωπαϊκών οδηγιών στην Ιταλία. Για παράδειγμα, λείπει ο ορισμός της έννοιας ευαλωτότητα. Συχνά δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μέτρα, να εφαρμόζονται δηλαδή, που προβλέπει η οδηγία και δεν υπάρχει ένα εθνικό ε, σχέδιο το οποίο πρέπει να εγκρίνεται ε, τρεις μήνες μετά την εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα το οποίο παρουσιάζει πολύ σοβαρά ελλείμματα. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερα τώρα με τις τεράστιες ε, περικοπές, ιδιαίτερα στο τομέα ε, αυτών. Η προστασία δηλαδή των θυμάτων πάσχει ε, μέσα από αυτή την πολιτική. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ όλο στην κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για αυτήν την έκθεση και πρέπει να πω ότι κανένας δεν ε, μπορεί να μην συγκινηθεί από αυτά τα ε, στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Ε, 80.000 άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, άντρες είναι σήματα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπορίες ανθρώπων και 60% και τις 100 από αυτούς προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν εγκληματικές δραστηριότητες αυτές αλλά δυστυχώς ε, πάρα πολύ προσοδοφόρες από επιχειρηματικής πλευράς. Θέλω να αναφέρω ξανά το θέμα των παιδιών, η πιο ευαίσθητη και βάλωτη ομάδα. Εκτός από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και διαβία εργασία, αυτό το οποίο σήμερα διαπιστώνουμε είναι μία νέα μορφή ε, εμπορίας ανθρώπων για αναπαραγωγικούς σκοπούς Δηλαδή, γυναίκες οι οποίες δέχονται να είναι έγκυες ε, ε, για παιδιά κατά παραγγελία ανάδοχες μητέρες και επίσης σε παιδιά που ε, γίνονται θύματα εμπορίας για υιοθεσίες. Υπάρχει λοιπόν ένας ολόκληρος τομέας, ένας τουρισμός που έχει δημιουργηθεί για την εξέβρεση ανάδοχων μητέρων. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πιστεύω πρέπει να προσθεθεί, δηλαδή εκμετάλλευση εμπορία ανθρώπων για αναπαραγωγικού σκοπούς. Η, Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά ευχαριστώ την δόκτωρα Βασιλιάδου για την ενεργητική και εμπεριστατωμένη ε, παρουσίασή της, τη δυναμική της παρουσίαση και εκ μέρους της κυρίας ε, Κέντριν Μπίρντα, η οποία είναι η άλλη ε, συντονίστρια, δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή της οδηγίας 2004 για την έκδοση αδειών παραμονής που ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων, Πώς θεωρείτε, πώς ε, αντιμετωπίζετε την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και τις συγκεκριμένες δράσεις προτείνετε ε, για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό των σημάτων αυτών και την συνειδητοποίηση από την πλευρά των σημάτων των δικαιωμάτων τους. Να καταλάβουν δηλαδή τι δικαιώματα έχουν δεδομένου ότι τα, οι άδειε παραμονής που έχουν εκδοθεί είναι πάρα πολύ λίγες και επίσης λαμβάνεται υπόψη στις διατάξεις αυτής της οδηγίας και στην εφαρμογή της η διάσταση των φύλων. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος, ο κύριος Κύρκος έχει το λόγο. Ευχαριστήσω την κυρία Βασιλιάδου για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά κυρίως για τα ερωτήματα τα οποία μας έθεσε και τις πολιτικές ερωτήσεις τις οποίες θα συναντήσουμε μπροστά μας και τις απαντήσεις θα πρέπει να τις ψάξουμε τα επόμενα χρόνια. Ήταν πραγματικά μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω μόνο και να ρωτήσω ε, στο θέμα των παιδιών τα οποία ε, ακολουθούν τα ρεύματα της μετανάστευσης, πάρα πολλές φορές χωρίς γονείς, βρίσκονται μόνα τους ε, στις χώρες μας, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ε, βρίσκονται σε ένα καθεστώς το οποίο είναι απροσδιόριστο. Ε, αν έχετε κάποια πολιτική απάντηση του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτά, εξειδικευμένα και όχι γενικότερα για το θέμα της μετανάστευσης. Thank you, Mr. Jurek. Ευχαριστώ κύριε Ντούρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ την ε, κυρία Βασιλιάδη για μια πάρα πολύ, για μια εξαιρετική έκθεση, διαφάνεια και εμπεριστατωμένη. Εγώ ξέρω ότι στην Πολωνία αστυνομικές ε, αρχές ε, ε, έχουν διαπιστώσει ότι τα όρια μεταξύ σεξουαλικής εκμετάλλευσης και παιδικής πορνείας και πορνογραφίας είναι πολύ ρευστά ε, όχι, λοιπόν, πρέπει λοιπόν να, να αντιμετωπίσουμε τα δικήματα αυτά, όχι μόνο να ποινικοποιήσουμε την χρησιμοποίηση των νόμων αυτών, τη δουλειά τους δηλαδή ότι είναι ποινικό αδίκημα, αλλά θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε και άλλες παράπλευρες δραστηριότητε όπως την πορνεία. Ε, στη Σουηδία, στη Γαλλία αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συζήτηση για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε εκμετάλλευση γυναίκας για κερδοσκοπία, για κερδοσκοπικούς σκοπούς ως αδίκημα ε, από κάποιον. Διαφορετικά δεν θα αντιμετωπίσουμε ε, αυτά τα φαινόμενα εδώ επισέχεται και το θέμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναλάβουμε παρόμοιες δράσεις. Ευχαριστώ κύριε Σουτζαντόσκι. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντονίστρια για αυτή την πολύ σαφή έκθεση. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για ένα πολύ συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο αναφέρατε. Ε, μιλήσατε για την ε, εργασία ε, ε, σε συνθήκες δουλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι που αφορά όχι μόνο πολίτες τρίτων χωρών, αλλά μερικές φορές και Ευρωπαίους πολίτες. Από χώρες της ε, κεντρικής Ευρώπης ή και της Ρουμανίας. Ή και τη Ρουμανία. Θα ήθελα να ρωτήσω τι συστήνεται, τι προτείνεται για αυτό το φαινόμενο. Είπατε ότι δυστυχώς η οδηγία δεν καλύπτει τους ε, εργοδότες οι οποίοι απασχολούν ε, άτομα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει μόνο θύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει, ότι είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η νομική κάλυψη. Έτσι ώστε να καλύπτονται και οι εργοδότες που απασχολούν θύματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω περιπτώσεις από την Ιταλία ή την κάτω χώρα, ίσως και υπάρχουν περιπτώσεις και σε άλλα κράτη-μέλη. πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καλυφθούν και αυτοί οι εργοδότες. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς τι θα θέλατε να γίνει. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Βαγίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βασιλιάδου για την ε, παρουσίασή σας. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, τι πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της ζήτησης για εμπορία ατόμων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Δεύτερον, ε, δεδομένου ότι γνωρίζουμε το πώς συνδέεται η εμπορία ανθρώπων με την πορνεία, τι, θα, τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν γι' αυτό. you, Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόνιμπολ. Um, Θέλω να σχολιάσω κάτι για το οποίο μίλησαν και προηγούμενοι ομιλητέ. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν την κυρία Βασιλιάδου για αυτή την πολύ σαφή παρουσίαση. Μα έδωσε καινούριε πληροφορίε. Ε, ε, μιλήσατε για την έκθεση περιπορνείας ε, και σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την ισότητα δύο φυλών. Είμαι εισηγήτρια για αυτήν την έκθεση, οπότε με ενδιαφέρει. κάτι για το, το οποίο αναφέρεται είναι ότι 65% των θυμάτων περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια και μιλάμε για ισότητα των δύο φύλων, όπως είπατε και εσείς, το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Έχουμε πλέον μια πολύ καλή βάση. Έχουμε την έκθεσή σας και άλλες εκθέσεις. Έχουμε αρκετά στοιχεία, αρκετή τεκμηρίωση. Επίσης έχουμε μιλήσει πολύ για τη μείωση της ζήτησης που παίζει ρόλο κλειδί. Η μείωση της ζήτησης σίγουρα θα μειώσει την εμπορία. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε γενικότερα τη σκέψη σας για το θέμα του φαινομένου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Χόνιβολ. Ολοκληρώνοντας δίνω το λόγο στην κυρία Μέγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έχουμε αναλάβει πολύ συχνά στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ε, η, πολιτική μετανάστευση και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσελκύει ε, ε, αυτό το φαινόμενο και το αυξάνει. Ακριβώς επειδή τα σύνορα μας είναι ανοιχτά. Πιστε, το πιστεύετε αυτό. Πιστεύετε ότι αυτή η πολιτική ε, προωθεί το φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Βασιλιάδου για να απαντήσει ε, αυτό τον πολύ ψηλό αριθμό ερωτήσεων. Ξέρω ότι είναι περιπλόκο, αλλά σας παρακαλώ πολύ, κυρία Βασιλιάδου, ε, να μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά, διότι έχουμε ακόμα ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν γίνεται να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα λεπτομερώς εδώ, ε, ίσως ε, θα μπορούσε αυτό να γίνει με άλλους τρόπους αργότερα άλλη στιγμή. Έχετε το λόγο κυρία Βασιλιάδου. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά το Κοινοβούλιο για όλο το ενδιαφέρον που δείχνει προκειμένου αυτό το θέμα να παραμείνει στην ημέρηση διάταξη των πολιτικών. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Να πω δύο λόγια μόνο. Πρώτον, πρόληψη ξεκινήσαμε μια ε, μελέτη για τις πρωτοβουλίες πρόληψης, γιατί η Κομισιόν έχει χρηματοδοτήσει με εκατομμύρια ευρώ ε, διάφορους, ε, οργανώσει οργανώσεις για την ευαισθητοποίηση, για την πρόληψη του φαινομένου κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι έχει δουλέψει και ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των εργασιών. Ξεκινάμε λοιπόν μια μελέτη για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ε, τη δουλειά που έχει γίνει και τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Θέλουμε πραγματικά όλες αυτές οι εργασίες να οδηγούν σε μείωση του αριθμού των θυμάτων. Ξεκίνησαμε λοιπόν αυτή τη μελέτη. Σε ό,τι αφορά την διαφορά ανάμεσα στο λαθρεμπόριο ανθρώπων και την εμπορία ανθρώπων. Όλοι συμφωνούμε. Ε, να υπογραμμίσω το εξή. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Εγώ πρέπει να τα υπερασπίσω, διότι πριν από τρία χρόνια όταν διορίστηκα γινόντουσαν πολύ λιγότερα πράγματα γιατί δεν υφίστατο η οδηγία, δεν υφίστατο η στρατηγική. Τώρα πια υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση, περισσότερη κινητοποίηση. Όμως και πάλι βρισκόμαστε στην αφετηρία. Γιατί η οδηγία είναι κάτι πολύ καινούριο, έτσι, υιοθετήθηκε πέρσι μόλις, ε, οπότε πρέπει να δούμε τα αποτελέσματά της. Και η έκθεση για την εφαρμογή της, όπως και η πρώτη έκθεση Ευρωπαϊκή Ένωσης για το τράφικινγκ του χρόνου, θα μας πούν πολύ περισσότερα πράγματα. Για συγκεκριμένα κράτη-μέλη δεν θα απαντήσω, αλλά μπορώ να σας πω ότι την Παρασκευή έληξε η προθεσμία και τα κράτη-μέλη υπέβαλαν τις εθνικές τους εκθέσεις προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε και να συντάξουμε την ευρωπαϊκή έκθεση τους επόμενους μήνες. Οπότε εκεί θα δείτε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε κράτος μέλος, τι έκανε το κάθε κράτος μέλος. Μιλήσατε επίση και για την κοινωνία των πολιτών και πολύ ορθά νομίζω. Να πω το εξή: έχουμε ενθαρρύνει και έχουμε εκφράσει την επιθυμία μας να συνεργαστούμε με την ε, κοινωνία των πολιτών. Οπότε η κοινωνία των πολιτών θα υποβάλει τις δικές της εκθέσεις, τα δικά της σχόλια ε, για το τι συμβαίνει στο επίπεδο του κάθε κράτους μέλους, ιδέες για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία και θα λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις συνεισφορές στη δική μας ευρωπαϊκή έκθεση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της συνένεσης. Το θέμα της συνένεσης δεν έχει καμία σχέση. Είτε πρόκειται για παιδιά, είτε πρόκειται για ενήλικους όταν μιλάμε για εμπορία ανθρώπων. Δεν τίθεται θέμα συνένεσης στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Γνωρίζουμε ότι εμπορία πολλές φορές γίνεται εντός μιας συγκεκριμένης κοινότητας ή ακόμα και εντός του οικογενειακού κύκλου του σογιού. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα παιδιά δίνουν, δεν δίνουν στη συνένεσή τους με επουδενή. Θα πρέπει ε, να διώκουμε τους ε, ε, υπετίους με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ας πούμε και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι μια οικογένεια πραγματικά εμπορεύεται τα παιδιά τους. Ε, ποιος ε, βγάζει το κέρδος, ε, προφανώς η ίδια οικογένεια. Αλλά ποιος ζητάει τις υπηρεσίες. Ποιος ζητά υπηρεσίες για την ε, εξεξουαλική εκμετάλλευση. Ε, ποιος τροφοδοτεί αυτό το, το σύστημα της επαιτίας στα φανάρια. Ε, αν κανένας, αν εγώ ήμουν παιδί που ζητούσα λεφτά στα φανάρια και κανένας δεν μου έδινε λεφτά, κανένας δεν ζητούσε τις υπηρεσίες μου, τότε το πρόβλημα θα άλλαζε. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά πιστεύω ότι τα περισσότερα παιδιά που επαιτούν στους δρόμους δεν είναι εκεί με τη μητέρα τους, είναι με άλλη γυναίκα. Ε, πολλά από αυτά τα παιδιά ε, εκβιάζονται και βιάζονται για να ε, επαιτήσουν. Ε, το εξετάζουμε το φαινόμενο, έχουμε μελέτη, έχουμε, τα ποσοστά είναι πολύ μικρά, αλλά ε, μιλάμε μόνο για τα καταγεγραμμένα θύματα. Ε, δεν υπάρχουν μόνο όμως καταγεγραμμένα θύματα, είναι πολύ μικρά, μικρός αριθμό των καταγεγραμμένων θυμάτων. Ε, το γνωρίζουμε αυτό και θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ περισσότερο το φαινόμενο. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο οργάνων. Χαίρομαι που το θέσατε το θέμα. Δεν είναι δυνατόν κανένα να μην γνωρίζει ότι υφίσταται αυτό το εμπόριο οργάνων. Κάποιοι γιατροί, κάποιοι ε, ε, εργαζόμενοι στις φαρμακευτικές εταιρείες το ξέρουν. Κάποιοι λοιπόν κλείνουν τα μάτια ή εν πάση περιπτώσει αν δεν το γνωρίζουν ε, κακώς δεν το γνωρίζουν. Και εκεί ε, μπαίνει στο παιχνίδι η εφαρμογή του νόμου. Αυτή τη στιγμή πλέον οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι υποχρεωμένες να γνωρίζουν ε, όταν απασχολούν θύματα εμπορίας. Μετά έχουμε νομοθεσία, έχουμε οδηγία ε, που ε, ε, διεθνείς έχουμε Συγγνώμη, έχουμε σε εθνικό επίπεδο νομοθεσία η οποία καταδικάζει τους εργοδότες που απασχολούν εγνώση τους θύματα trafficking αλλά δεν το έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, θα υποβάλουμε προτάσεις. Το 2016 το έχουμε αναλάβει να το κάνουμε, αλλά το 2016 είναι αύριο. Τώρα, ε, για την, ε, τη ζήτηση. Το επαναλαμβάνω συνεχώς. Πρόκειται για θέμα ζήτησης. Ε, πρόκειται για λεφτά. Ε, όχι μόνο για τους παράνομους τομείς, αλλά και στους νόμιμους τομείς οικονομίας που βγάζουν χρήματα από το, την εμπορία. Αν είχαμε μόνο τους παράνομους εμπόρους, ε, θα είχαμε λιγότερα προβλήματα. Όπως είπατε και εσείς, λαμβάνουμε υπόψη πολύ το θέμα της ζήτησης. Έχουμε ξεκινήσει επίσης μια μελέτη για το φύλλο, ε, για την ποινικοποίηση αυτών που εν γνώση τους κάνουν χρήση υπηρεσιών θυμάτων και θα συνεχίσουμε, αν χρειαστεί, με προτάσεις με βάση τα πορίσματά μας. Μπορώ να πω κάτι τώρα, όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά μπορώ να σας πω ότι το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Υφίσταται αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνθήκη, σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς επίσης και την εκμετάλλευση της πορνείας άλλων. Και όπως είπαν πολλοί βουλευτές, ε, αυτή η πορνεία είναι ένας τομέας ψηλού κινδύνου. Ε, πρόσφατα κάποιος υπεύθυνος της ε, γερμανικής αστυνομίας είπε ε, ότι ε, όλα τα θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ήταν στο κύκλωμα της πορνείας. αυτό ίσως δεν είναι ο απόλυτος κανόνας, θα πρέπει να, τις, τα προστατεύσουμε. Τώρα, για τα, βάλω τα παιδιά και τους ανήλικους. χρειάζονται συστήματα προστασίας των παιδιών. Τα παιδιά είναι παιδιά καταρχήν ανεξαρτήτως του στάτους τους και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, ποια είναι η ηλικία και τη ομάδα κλπ. Καταρχήν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως παιδιά, ανεξαρτήτως του στάτους τους. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε το, σύστημα, το θέμα της, ε, των συστημάτων προστασία των παιδιών. Και τέλος, ασφαλώς θα πρέπει να συνδέσουμε το θέμα αυτό με την πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Το καταλαβαίνω. Πρέπει όμως να πω ότι μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Οπότε δεν πρόκειται μόνο για θέμα μετανάστευσης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τους προστατεύσουμε από, το, από τη θυματοποίησή τους. Και βέβαια θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τα λεφτά. Follow the money. Follow the money σε όλα τα κυκλώματα, σε όλους τους τομείς. Ποιος ωφελείται, εν γνώση του ή ε, εναγνία του, από αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει να δούμε πού πάει το χρήμα σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς που συνδέονται με αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Dr. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Βασιλιάδου. Από το χειροκρότημα βλέπετε ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Ο χρόνος μας πιέζει. Θέλουμε όμως ε, να προχωρήσουμε. Ε, η οδηγία του 2011 δημιούργησε ένα συντονισμό μεταξύ πολλών οδηγιών και σύνθετων θεμάτων. Δεν μπορέσαμε σε ένα πρωινό να καλύψουμε τα πάντα. Μας είπατε όμως ε, όσα περισσότερα γινόταν πρέπει να πω. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πολλά από αυτά τα θέματα. Όμως ε, σας παρακαλώ να σημειώσετε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και η πρόεδρος της Επιτροπής ΦΑΜ που είπε ότι Χρειαζόμαστε περισσότερη συμβολή από τα μέλη μας και θα αναζητήσουμε ευκαιρίες για να γίνει αυτό. Διότι και τα νέα μέλη θέλουν, ε, θα θέλουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι αναφέραμε σήμερα, γιατί τα θέματα είναι πολύ περίπλοκα. Και κάποιοι εισηγητές επίσης θέλουν και να συμβάλλουν και να ενημερωθούν. Ε, ε επιφανειακά το καταπιαστήκαμε το θέμα σήμερα το πρωί, γιατί είναι δύσκολο. Ε, βέβαια δεν θα σας ε, δώσω πέντε ώρες, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο. Ίσως ε, θα πρέπει να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος ε, πιάνοντας τα επιμέρους μέρη αυτού του θέματος. Σας ευχαριστούμε και ελπίζω να σας ξαναδούμε πολύ γρήγορα. Ζητώ συγγνώμη από την επόμενη προσκεκλημένη μας, την ε, κυρία Κριστίνα Κάγκας Πούντα, η οποία είναι από τα Ηνωμένα Έθνη. Έρχεται. Γρήγορα ελπίζω να έρθει, γιατί ο χρόνος μας πιέζει πολύ. Ωραία. Η εμπορία είναι παγκόσμιο θέμα Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και στην προσκεκλημένη μας και όλους σας που τόσο πολύ πιέζω ε, στην ημερήσια διάταξη. Ήταν αναπόφευκτο βέβαια να δώσουμε περισσότερο χρόνο σήμερα το πρωί στη συντονίστρια. Η κυρία Καγκασπούντου είναι επικεφαλής ε, της ε, μονάδας ε, υπεύθυνη για την Παγκόσμια Έκθεση για την Εμπορία Ανθρώπων στο στο Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκλήματος. Είναι παγκόσμιο θέμα, εδώ έχουμε και έμπειρα μέλη που γνωρίζουν και ε, τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να παρουσιάσουμε εν συντομία το θέμα, να δούμε τι ερωτήσεις υπάρχουν και αν είναι λίγες οι ερωτήσεις μπορείτε να προσθέσετε στην πρώτη συνοπτική σας παρουσίαση. Συγγνώμη και πάλι που σας πιέζω και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω εδώ. Έχω μια ε, παρουσίαση PowerPoint που θα τη δείξω πολύ γρήγορα, δεν ε, είναι, πολύ σύντομη, καταλαβαίνω ότι έχετε χρονικές πιέσεις. Να πω επίσης ε, ότι νιώθω λίγο ξένη εδώ, είμαι από τον ΟΗΕ, είναι, με ξενίζει λίγο το περιβάλλον. Ε, όλοι ξένοι είμαστε, λέει ο πρόεδρος, εδώ. εντάξει, αλλά τα οργανωτικά σας δεν τα γνωρίζω πολύ καλά. Εσείς μιλάτε για την εμπορία ανθρώπων, εμείς μιλάμε για εμπορία προσώπων. Θα μιλήσω λοιπόν με αυτή την ορολογία γιατί αυτήν έχω συνηθίσει. Το Γραφείο για τα Ναρκωτικά και του Εγκλήματος του ΟΗΕ έχει εδώ και χρόνια παρουσιάσει εκθέσεις, η τέταρτη είναι αυτή που η έκθεση και έχουμε τέσσερα μέρη, το ένα το πιο λεπτό είναι οι παγκόσμιες και οι περιφερειακές, περιφερειακές πρόπτικες και το πιο μεγάλο κομμάτι υπησέρχεται στο προφίλ των χωρών που καλύψαμε στην έκθεση. 158 χώρες καλύφθηκαν στην έκθεση αυτή την τέταρτη και το προφίλ των χωρών, δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Εδώ βλέπετε την κάλυψη της παγκόσμιας έκθεσης και τις χώρες που δεν ανταποκρίθηκαν και δεν απάντησαν σε ερωτήσεις. Οι χώρες αυτές συνήθως βρίσκονται στην Αφρική και την Ασία. Τώρα, κάποια βασικά μας ευρήματα με βάση την ανάλυση των δεδομένων που κάναμε. Καταρχήν, η διακίνηση ανθρώπων γίνεται παντού. Τα θύματα προέρχονται από 152 χώρες 152 ε, διαφορετικές ε, ηθαγένειες υπάρχουν από 124 χώρες το 2010-2012. Επίσης διαπιστώσαμε ότι ε, εντοπίσαμε 510 ροές εμπορίας ατόμων, δηλαδή 5 άτομα από το, τουλάχιστον από, τον ίδιο από την ίδια προέλευση, τον ίδιο προορισμό. Και Υποθέτω ότι δεν καλύψαμε και όλες τις χώρες, μπορούμε με αρκετή ασφάλεια να πούμε ότι όλες οι χώρες έχουν κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, οι ροές που εντοπίσαμε, τα ρεύματα. Έχουμε υπερεθνικές ε, ροές, δηλαδή ταξιδεύουν, διακινούνται μεταξύ υπήρων. Ε, ένα είναι από τη Μέση Ανατολή, α, ε, ως σημείο προορισμού. Το άλλο είναι η Βόρεια Αμερική και η Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική και η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Και βλέπετε ότι η βασική προέλευση για αυτούς τους προορισμούς είναι η Ποσαχάρη Αφρική, η Νότια Αμερική, Νότια Ασία και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, οι ροές είναι από τις πτωχές στις πλούσιες περιφέρειες και το είδαμε αυτό και σε περιφερειακή βάση και σε βάση χωρών αναχώρα. Η εμπορία ανθρώπων είναι υπερεθνικό ε, έγκλημα, αξιόπινη πράξη που ε, ενέχει πολλές φορές και εγχώριους παραβάτες και έχει περιορισμένη εμβέλεια γεωγραφική. Βλέπετε εδώ συνήθως υπάρχει κίνηση στην υποπεριφέρεια. Το 34% είναι σε εγχώριο επίπεδο, σε μια χώρα, τα υπόλοιπα είναι ε, υπερεθνικά, διασυνοριακές δηλαδή διακινήσεις. Υπέρ τα περισσότερα θύματα που εντοπίζουμε είναι αλλοδαπή αλλά οι περισσότεροι διακινούνται υποπεριφερειακά, γιατί μόνο ένα τέταρτο των θυμάτων εμπορίας ε, πάνε μεταξύ υπήρων, διακινούνται μεταξύ υπήρων ή περιοχών, περιφερειών. Επίσης, οι περισσότεροι διακινητές που εντοπίζονται, που είναι οι δράστες, ε, οι εγκληματίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν καταδικαστεί. 64% των καταδικασμένων διακινητών είναι ε, υπήκοοι της χώρας όπου καταδικάστηκαν. Υπάρχουν και κάποια ποσοστά αλλοδαπών από την ίδια περιφέρεια ή από άλλες περιφέρειες που ε, καταδικάστηκαν στις χώρες αυτές. Επίσης υπάρχει αυξημένος εντοπισμός διακίνησης για στόχους άλλους εκτός από την σεξουαλική εκμετάλλευση. Η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι η βασική μορφή εκμετάλλευσης ε, της, στην εμπορία. 53% περίπου είναι ε, θύματα τέτοιας εκμετάλλευσης, 40% παγκοσμίως των θυμάτων έχουν ε, καταναγκαστική εργασία και κάποιες άλλες μορφές 7%. Το ε, ε, συνεχές έβριμα είναι ότι τα θύματα καταναγκαστικής εργασίας έχουν αυξηθεί. Αυτό ε, δηλαδή ο εξαναγκασμός σε εργασία δεν εντοπίζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περιφέρεια αυτή, παρόλο που αυξάνεται σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Και αυτό το δείχνει και αυτή η σύγκριση περιφερειών. Βλέπετε στην Ευρώπη που είναι με κόκκινο χρώμα, που, όχι, η τελευταία, τελευταία σειρά και με κόκκινο φαίνεται η σεξουαλική εκμετάλλευση σε ποσοστό 66% των θυμάτων λοιπόν είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, 26% καταναγκαστική εργασία. Αν τα συγκρίνουμε αυτά με την Ανατολική Ασία, Νότια Ασία και τον Ειρηνικό, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, διότι σε αυτή την περιφέρεια το 64% των θυμάτων ε, πάνε για ε, εξαναγκασμό σε εργασία. Διαφέρουν τα ποσοστά λοιπόν ανάλογα με την περιφέρεια όπως βλέπετε. Επίσης οι γυναίκες συμμετέχουν πάρα πολύ στην εμπορία ανθρώπων και ως θύματα και ως παραβάτες περίπου το 30% των διακινητών που εντοπίζονται είναι γυναίκες, πολύ υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες αδικοπραξίες όπου το ποσοστό των καταδικασμένων γυναικών είναι από 10 μέχρι 15%. Τούτο εδώ είναι κατ' πολύ ψηλό. Επίσης, ε, ε, βλέπουμε τα θύματα εδώ περίπου 50% των γυναικών, ε, θυμάτων είναι γυναίκες, ε, κορίτσια κάτω από 18 είναι 21%. Αν τα προσθέσουμε πάμε στο 70% δηλαδή ε, γυναίκες και κορίτσια και έχουμε και ενήλικους άνδρες και αγόρια. Αν δούμε επίσης ε, τη το 70% των γυναικών θυμάτων, οι περισσότερες ε, πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αν δούμε παγκοσμίω όμως την ομάδα εκείνων που ε, ε, έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης για εξαναγκασμό σε, βλέπουμε, σε εργασία, βλέπουμε 35% των θυμάτων είναι γυναίκες. Οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ενώ οι άνδρες πάνε κυρίως για ε, εξαναγκασμό σε εργασία, οι γυναίκες ε, πέφτουν θύματα και εξαναγκασμού σε εργασία και ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Είπα πολλές φορές ότι αυξάνεται η εμπορία παιδιών που εντοπίζεται, εδώ βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα με πράσινο χρώμα τα, τις περιπτώσεις κοριτσιών θυμάτων που εντοπίζονται και όπως βλέπετε τα προηγούμενα 10 χρόνια το ποσοστό των κοριτσιών θυμάτων αυξήθηκε από το 10% στο 21% και αυτό το βλέπουμε να είναι πολύ ανησυχητικό, πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε πολύ μεγάλες περιφερειακές διαφορές στην Ευρώπη και Κεντρική Ασία 18% των, ε, των ε, θυμάτων είναι κορίτσια. Αν δούμε την Αφρική, η Ποσαχάρη Αφρική, πάνω από 60% των θυμάτων εδώ είναι παιδιά. Αν δούμε την ομοθεσία και την ποινικοποίηση, βλέπουμε ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν καλύπτονται όπως πρέπει ε, με βάση το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ε, προσώπων, ε, το οποίο το 2003 τέθηκε σε ισχύ και μετά, αν δούμε την κατάσταση ως προς την νομοθεσία, βλέπουμε ότι μόνο 9 χώρες, το 5% των χωρών δηλαδή, δεν έχουν καμία απολύτως νομοθεσία για αυτό το θέμα. Και άλλο ένα 10% ε, των χωρών έχουν μόνο εν μέρη νομοθεσία. Σημαίνει δηλαδή ότι μέρος μόνο ε, των ε, μπόρων προσώπων ποινικοποιείται. Καλύπτονται μόνο κάποια θύματα και όχι όλα αν υπολογίσω με τον πληθυσμό αυτών των ανθρώπων που έχουν μόνο μερική νομοθεσία ή που δεν έχουν καθόλου σχετική νομοθεσία, πάμε σε, στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που είναι πάρα πολλοί. Όμως, αν είχαμε επιτυχία με την νομοθεσία μας, δεν είχαμε με τις ε, καταδίκες μεγάλη επιτυχία και κυριαρχή η ατιμορρησία. 50 ε, χώρες δεν είχαν έχουμε 26% χωρών που είχαν λιγότερες από 10 καταδίκες. Και τα κακά νέα είναι ότι η κατάσταση δεν άλλαξε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Έχει σταθεροποιηθεί και δεν αυξάνεται ο αριθμό των καταδικών. Σταματώ εδώ. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας η έκθεση και βεβαίως Ευχαριστώ να σας στείλω και το έγγραφο αν χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ασφαλώς θα θέλατε να πείτε περισσότερο γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο θέμα και μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες. Ξέρουμε λοιπόν την μεγάλη σημασία αυτής της έκθεσης. Σα κάτσουν διερμηνείς ε, λίγο περισσότερο ε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε δύο-τρεις ερωτήσεις και να απαντήσει η ομιλήτρια. Από ό,τι βλέπω όμως δεν υπάρχει καμία ερώτηση. Α. Ε, ευχαριστώ ε, την ε, ομιλήτρια για την παρουσίασή της. Έχω δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, ξαναρχίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Η πρώτη μου ερώτηση είναι εάν καλύψατε και το βιομηχανικό τομέα και τις βιομηχανίες τις οποίες εργάζονται ή απασχολούνται τα σήματα και δεύτερον διαπιστώνουμε τον αυξημένο αριθμό παιδιών που υποχρεώνονται να, να, συμμετέχουν σε πολέμους. Είναι πάρα πολύ μικρά παιδιά αυτά, τα οποία διαβίες εξαναγκάζονται να, να πάρουν όπλα και να πολεμήσουν. Έχετε στοιχεία? Ο πρόεδρος. θα πρότεινα να ανταλλάξετε στατιστικές ε, πληροφορίες ε, με τον συντονιστή μας ε, και θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχουν στατιστικά κενά ή στατιστικά προβλήματα στην διαδικτυακή συνεργασία με, τον, με τη δική μας συντονίστρια Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ερώτηση ενδιαφέρουσα και αν μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές και ευχαριστώ τους διερμηνείς, θα παραμείνει λίγο λεπτά ακόμα, λέει ο Πρόεδρος. Ε, εάν κατάλαβα καλά την ερώτηση, αναφερθήκατε στην ε, ε, διαβίαση, αναγκαστική εργασία σε βιομηχανικό τομέα και για τα παιδιά στρατιώτες πραγματικά είναι ένα πολύ ανισχυτικό αριθμό παιδιών τα οποία έχουν εξαναγκαστεί να πολεμήσουν και έχουν διακινηθεί για ακριβώς αυτή την συμμετοχή τους σε διάφορες ένοπλες ομάδες αυτές τις ε, περιοχές σειράξεων. Όχι μόνο χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά στρατιώτες, αλλά τα εκμεταλλεύονται και σεξουαλικά και με άλλες μορφές. Έχουμε λοιπόν πραγματικά πληροφορίες για αυτό το θέμα και η κατάσταση είναι κακή. Όσον αφορά για την, τον εξαναγκασμό σε εργασία, ε, εννοείται εξαναγκαστική εργασία και άλλες μορφές διακίνησης ατόμων, ανθρώπων, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαφορετικές μορφές εξαναγκαστικής εργασίας, αναγκαστικής εργασία. δυστυχώς δεν έχουν καταγραφεί όλες αυτές οι μορφές γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία σε πολλές χώρες και δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ε, ορισμός ε, για τις εργασίες αυτές και πολλές φορές διαφεύγει η καταγραφή τους ως εξαναγκασμός σε εργασία. Ε, πάντως, όποτε είναι δυνατόν πρέπει να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη κατά αυτών εργοδοτών και υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων για την συνεργασία με το όργανο, με το φορέα ε, κατά της ε, ε, διακίνησης εμπορίας ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, μια εξαιρετική ευκαιρία όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνουμε την ε, ευρωπαϊκή, συμπληρώνουμε την παγκόσμια εικόνα που έχουμε για το θέμα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία και αντίστροφα. Ε, πολλές φορές τα στοιχεία αυτά είναι διαπεριφερειακά και καλύπτουν μεγάλες περιοχές του κόσμου και πολλές φορές είναι, ε, διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες 130 χωρών από 130 διαφορετικές χώρες ταυτοποιήθηκαν ως θύματα στην Ευρώπη. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός διαφορετικών εθνικοτήτων, σημάτων και ενώ μιλάμε ε, για τα ίδια θέματα, φαινόμενα, στοιχεία και προβλήματα, υπάρχουν ορισμένα ορισμένες μικρές διαφοροποίησεις μεταξύ των περιπτώσεων ανάλογα με την προέλευσή τους και μπορούμε σαφώς να συνεργαστούμε σε βάθος σε αυτό το θέμα. Ο Πρόεδρος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Συνάδελφοι, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις και εκ μέρους των δύο ε, επιτροπών, ε, λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.